μία δεύτερη παρατηρήση, μία δεύτερη ανακοίνωση και μία τρίτη. Σύμφωνα με τα άρθρα του κώδικα δεοντολογίας στις 25 Νοεμβρίου 2014 αποφασιστικά τώρα του Τζον Μαρί Καβαντά ως μέλο της Συμβουλευτικής Επιτροπής ε, για την συμπεριφορά των μέλων να τον ορίσω στη θέση του κυρίου Σώσα Βάγνα. Και η τρίτη ανακοίνωση από την ομάδα των φιλελευθέρων ε, έλαβα αιτήματα για διορισμούς σε επιτροπές και ε, αντιπροσωπείες. Ο κατάλογος των προτινόμενων θα δημοσιευθεί